για την κοινωνική δράση σε σχέση με την φαλαινοθυρία. Ορμαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Αουτούλ. Ακολουθεί η έκθεση του κυρίου Μπέλετ για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικού. Ονομαστική ψήφος, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην, στον εισηγητή μας. Ακολουθεί η έκθεση του κυρίου Φάβα για τις κυρώσεις εναντίον αυτών που απασχολούν παράνομους ε, πολίτες τριτών χωρών. Έχουμε το νομοθετικό ψήφισμα χωρίς τροπολογίες ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Φάβα. Ακολουθεί η έκθεση της κυρίας Γιεγκλ για τις στατιστικές αγροτικών προϊόντων. Ψηφίζουμε την πρόταση κανονισμού. Έχουμε δύο ομάδες τροπολογιών. Πρώτο μπλοκ θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία στο μπλοκ 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η πρόταση Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί ψήφι Κατά. Άποχες. Ενεκρίθη. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης. Συγχαίρω την εισηγητριά μας. Ακολουθεί η έκθεση του κυρίου Σάιερ για τους αρωματικούς ίνους. Ψηφίζουμε την πρόταση κανονισμού. Έχουμε δύο ομάδες τροπολογιών. Πρώτο μπλοκ, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ψηφίζουμε ψηφιπέ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η πρώτη ομάδα τροπολογιών. Η πρόταση της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Σάγερ ακολουθεί η έκθεση Βαντεμπύρχ για το, τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ψηφίζουμε την πρόταση οδηγίας. 7 χωριστές τροπολογίες. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 1. Παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Όλα αυτά είναι πολύ συναρπαστικά, λέει η Προεδρεύουσα. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω απορρίπτεται σαφώς αγαπητοί συνάδελφοι αν θέλετε εντάξει ψηφοφορία επαλήθευση για τροπολογία παριθμών 2 ψηφίσατε όλοι έληξε η ψηφοφορία και νεκρήθη. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και πάλι. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Μήπως είναι της Λούλινγκ αυτή. <laughs> Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για την 5 θα κάνουμε κατευθείαν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γιατί είναι μικρές οι διαφορές. Τροπολογία 5, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά την 5 η τροπολογία 4 πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. <clears throat> Τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε ψη, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και το νομοθετικό ψήφισμα <clears throat> με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Ακολουθεί το θέμα τεσσάρων ψηφισμάτων για την καταγγελόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη ΣΥΑ για την κράτηση και παράνομη μεταφορά κρατουμένων. Θα ψηφίσουμε ένα κοινό σχέδιο ψηφίσματος από τέσσερις πολιτικές ομάδες. Έχουμε λοιπόν την τροπολογική απεριθμών 1, την οποία θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Έναξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα το εκτιμώντας Β, Παύλα 4, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν τώρα στο εκτιμώντας Β, Παύλα 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορία ηλεκτρονικής παρακαλώ. Για το εκτιμώντας Β, Παύλα 5. Έναρξη. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. να ψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα στο σύνολό του, σε ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη, παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, το επόμενο είναι η έκθεση του κυρίου Σαρουσβάλσκι για την ετήσια έκθεση για τις βασικές πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΑ. Ψήφισμα, σχέδιο ψηφίσματος ψηφίζουμε. Καταρχάς η τροπολογία 9, υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η 8, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαρθμών 5 με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 και αυτή με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Αν ψήφισατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 1. Να δούμε ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Υπέρ της τροπολογίας 1. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 4 και 7 που είναι ταυτόσημες. Ονομαστικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 10 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ηλεκτρονικά να ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία για την 10, την τροπολογία υπαριθμών 10. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. το σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνάμε τώρα, μάλλον να κάνουμε ένα διάλειμμα στις ψηφοφορίες μας και θα συνεχίσουμε αργότερα.